La Presidente. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίαση και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί έχουν διανεμηθεί. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσει ή αντιρρήσει. τα πρακτικά θεωρούνται ότι έχουν